Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίασης είναι διαθέσιμη. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να παρέμβει. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο στην